Great. So, Mr. Saliba, if you can hear us, thank you for giving us the evidence. Λοιπόν, κύριε Σαλίβα, να μας ε, ακούσετε πολύ ωραία, μπορούμε να ξεκινήσουμε νομίζω. Έχετε το λόγο για την παρουσίαση του σχεδίου έκθεσή σας. Καλό απόγευμα και συγγνώμη που δεν μπορούσα να συνδεθώ. το σχέδιο έκθεση θέλει να βρει λύσεις. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ κακός ο ήχος και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον ομιλητή, οπότε θα λέμε ότι μπορούμε. Η έκθεση αυτή αναγνωρίζει ότι η ψηφιοποίηση έχει πολλά πλεονεκτήματα και για του εργοδότε και για του εργαζόμενου, μέχρι των οποίων και η ευελιξία. Η ευελιξία είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο προσφέρει μεγαλύτερη αυτονομία, μειώνεται ο χρόνος ε, αναμονής, από την άλλη ε, μπαίνουμε σε μια κουλτούρα που είμαστε συνέχεια συνδεδεμένοι. Τα θεμελιώδη δικαιώματα διακυβεύονται, ακόμα και οι δίκαιοι και οι ε, θεμητοί, εν πάση περιπτώσει, και αξιοπρεπής αμοιβή. Από την αρχή του COVID-19 και της πανδημίας, οι ευέλικτες ε, συνθήκες εργασίας ε, από απόσταση έχουν αποδειχθεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις, για κάποιες βιομηχανίες. Είχε αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων που τηλεργάζεται και ε, ενδέχεται να συνεχιστεί να, να χρησιμοποιείται αυτή η μέθοδος εργασίας και μετά την πανδημία. Βεβαίως υπάρχουν και κίνδυνοι, υπάρχουν και απειλές για τους εργαζόμενους. Διότι έχουμε συνθήκες εργασίας, ώρες εργασίας μακροσκελής και αυξημένες απαιτήσεις. Πιο μακροπρόθεσμα λοιπόν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα αυτά και είναι κάτι που επήγει. Υπάρχει πρόβλημα με τις ώρες εργασίας, με τις εβδομάδες εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν δικτύες ασφαλείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας για τους εργαζόμενους σε αυτό, τον το νέο τρόπο εργασίας. Έτσι λοιπόν χρειάζεται μια οδηγία για το δικαίωμα αποσύνδεσης. Αυτά είναι κάποια τα βασικά στοιχεία του σχεδίου έκθεσης. Πρώτα απ' όλα, η αποσύνδεση θα πρέπει να είναι ένα δικαίωμα, να περιγράφεται επακριβώς ως δικαίωμα των εργαζομένων, χωρίς κανένα ψηφιακό εργαλείο δηλαδή, να μην απαντούν για ένα διάστημα σε mail, σε τηλέφωνα, σε SMS, χωρίς να έχουν καμία επίπτωση εργασιακή. Αυτό πρέπει να αφορά όλους τους εργαζομένους, χωρίς, κανένα, ε, χωρίς καμία διάκριση. Για όσους χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία στη δουλειά τους, σε όλους τους τομείς δραστηριότητα και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Το δικαίωμα αποσύνδεση βασίζεται στο άρθρο 153 της συνθήκης ιδιαίτερα τα σημεία αβ παράγραφος 1. Πρέπει να είναι δίκαιες οι συνθήκες εργασίας, δίκαιη η αμοιβή και βεβαίως να υπάρχουν και όλες οι κατάλληλες, ε, όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις και όροι εργασίας ό,τι αφορά τις άδειες σεβασμός, απόλυτος σεβασμός της νομοθεσίας περί, περί εργασίας πρακτικοί διακανονισμοί για την εφαρμογή του δικαιώματος της αποσύνδεσης πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συμφωνίες μεταξύ των κοινωνικών εταίρων μέσω συλλογικών συμφωνιών μεταξύ εργοτών και εργαζομένων. Ένα από τα πιο βασικά άρθρα της οδηγίας που προωθούμε αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο που παίζουν οι κοινωνικοί εταίροι σε αυτή τη διαδικασία και βεβαίως θα πρέπει η εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε κλάδου και τις ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου και τις κάθε περιοχές, περιοχής και περιφέρειας. Αυτό που θέλουμε είναι να εξασφαλίσουμε ότι κάποιες οι προϋποθέσεις για το δικαίωμα αποσύνδεσης θα αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας, μέτρα για να μπορεί κάποιο να αποσυνδέεται τελείως από τα ψηφιακά εργαλεία, χωρίς παρακολούθηση να υπάρχει μια αξιολόγηση επίσης της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων όταν δουλεύουν σε ψηφιακό περιβάλλον και πρέπει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και αναπερίπτωση να προβλέπονται εξαιρέσεις. Πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε μια επιπλέον αποζημίωση κάποιων που εργάζεται πέρα των ορών που προβλέπονται. Οι εργοδότες θα πρέπει να δώσουν στους εργαζόμενους γραπτές πληροφορίες για τις, τις διατάξεις της συλλογικής αυτής συμφωνίας ό,τι αφορά την εφαρμογή του δικαιώματος αποσύνδεσης και για τη μέθοδο που θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να υποστηριχθεί αυτό το δικαίωμα. Επίσης, υπάρχει μια πρόταση για την διασφάλιση των εργαζομένων για να μην υπάρξει θυματοποίηση ή αρνητικές επιπτώσεις για τους εργαζόμενους που ασκούν το δικαίωμά τους και να μπορεί να υπάρχει και μια δυνατότητα προσφυγής όταν δεν εφαρμόζονται οι σωστές προϋποθέσεις. Δεν έχει νόημα να έχουμε μια καλή νομοθεσία όταν δεν είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε τις ασφαλεία ασφαλείας που θα επιτρέψουν την εφαρμογή της. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της πρότασης. Περιμένουμε με ανυπομονησία να συνεργαστώ με τους κοιόδης συζητητές για αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον και σημαντικό φάκελο και ελπίζω να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο φιλοδοξίας και να κάνουμε τη διαφορά για τη ζωή εκατομμυρίων εργαζόμενων, εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρουσίαση και τώρα περνάμε στους κοιόδης εισηγητές και τους εκπροσώπους των κομμάτων από το ΕΛΚ και η κυρία δεν είναι εδώ όμως. Συνεχίζουμε με τη Renew, κυρία From, ούτε αυτή είναι συνδεδεμένη. Η κυρία Λίτση για την ID είναι συνδεδεμένη. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Για δύο λεπτά. Λίτση, you have the floor. Α, να είμαστε. Καλημέρα. Γεια σας, συνάδελφοι, όσοι είστε συνδεδεμένοι, κύριε ε, εισηγητά, κυρία Πρόεδρε, πρέπει να σας διευκνήσω ότι σήμερα μπορέσαμε να ψηφίσουμε γιατί οι συνάδελφοι του ED είμαστε εδώ, κάναμε τη δουλειά μας και έτσι δώσαμε τη δυνατότητα στο να γίνει ψηφοφορία αυτό να μην ξεχαστεί. Όσον αφορά το θέμα μας πρέπει να σας πω ότι αυτή η σημαντική αύξηση στη χρήση αυτών των ε, εργαλείων ε, όσον αφορά ε, κάποιους καινούριου τρόπους εργασίας, όσον αφορά ε, διάφορε πτυχέ εργασίας, ιδίως όσον αφορά επίσης την αύξηση της τηλεργασία λόγω της πανδημίας, ανέδειξε το πρόβλημα. Θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες εγγυήσει για τους εργαζομένους, ούτω ώστε να ανακατοχυρθεί το δικαίωμα τη αποσύνδεση για να μην βλαβεί η υγεία του και η ευημερία τους γενικότερα. Να σας πω τώρα ε, ε, κάποια θέματα που με προβληματίζουν. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να βρούμε κάποιες πρακτικές λεπτομέρειες. Πώς δηλαδή θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε με συγκεκριμένο τρόπο αυτό το δικαίωμα. Είναι το θέμα της προστασίας ιδιωτικού βίου. Έχει κοπεί ο ήχος της κυρίας Λίτση. Ξανασυνδέεται κυρία Λίτση. Άρα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις εγγυήσεις που πρέπει να υπάρχουν ε, ε, για τους εργαζομένους, δηλαδή να υπάρχει κάποιο είδους ενημέρωση, κατάρτιση του εργαζομένου με κάποιον τρόπο ε, για, αυτό που περνάνε. Ξανακόβεται η κυρία Λίτση. Να δούμε τι γίνεται και με τις ε, γυναίκες. Αν υπάρξει κάποια παρέκκληση για το δικαίωμα της αποσύνδεσης θα πρέπει να καθοριστούν τα κριτήρια Πώς δηλαδή θα υπάρξει κάποια αντιστάθμιση χρηματική. Όσον αφορά δε τις γυναίκες, ακριβώς επειδή είναι κατάσταση τώρα πολύ εξαιρετικών συνθήκων, θα πρέπει να δούμε πώς θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες διότι η κατάστασή τους που ήδη είναι δύσκολη θα γίνει ακόμα χειρότερη και τι θα πρέπει να δούμε ότι οι γυναίκες πρέπει να φροντίσουν τα παιδιά. Στο έγγραφο της έκθεσης, στο σχέδιο του κειμένου, δεν αναφέρεται τίποτε για αυτό το πρόβλημα. you information Ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία Σάντερ, για το ΕΛΚ έχει ζητήσει να πάρει το λόγο, οπότε σας ερωτώ, ε, θέλετε να πάρετε το λόγο εκ μέρους της κυρίας Δεχόσκη, η οποία είναι σκιώδης συζητής εκ μέρους του ΕΛΚ ή εσείς θέλετε για σας την ίδια να πάρετε το λόγο. Κυρία Σάντερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να αντικαταστήσω τον σκιώδη συγητή, θα σας τα πω ε, τα θέματα τα δικά μου προσωπικά. Ε, σε αυτή την περίπτωση θα λάβετε το λόγο, αλλά αφού ολοκληρωθεί ο γύρος απόψεων των σκιωδών. Κυρία Ντεσούτο, των Πρασίνων. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή για την εξαιρετική του δουλειά μέχρι τώρα, ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη ε, και την πρόσφατη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Ε, πραγματικά και εγώ συμφωνώ με κάτι το οποίο έχει υποστηρίξει εδώ και πολύ καιρό η δική μου πολιτική ομάδα σε ό,τι αφορά την. Ε, μείωση του χρόνου εργασίας. Ε, στα σημεία 3 και 15 αναφέρεται ε, και κάτι τέτοιο βέβαια θα μπορούσε να βοηθήσει και στη διατήρηση των θέσεων εργασία. Τώρα τα όσα συνέβησαν πρόσφατα είναι πρωτόγνωρα. Έχουμε δηλαδή μεγαλύτερο χρόνο εργασίας, περισσότερες ώρες εργασίας και όχι τόσο τακτικέ. Αυτό το είδαμε ειδικότερα στο πλαίσιο της τηλεεργασία λόγω της κρίσης του COVID και βέβαια αυτό με τη σειρά του έχει επιπτώσεις στην φυσική αλλά και στην ε, ψυχική υγεία. Αυτό που θα ήθελα να ε, ζητήσω από τον εισηγητή να συμπεριλάβει κάποια δεδομένα από την ε, τελευταία έρευνα σε ό,τι αφορά την εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε ενδεχομένω θα μπορούσε να συμπεριλάβει κάποια τέτοια δεδομένα. Επίση, μια άλλη πρότασή μα είναι να ενισχυθούν λίγο περισσότερο οι πτυχέ που αφορούν στην ισότητα των φύλων μέσα στην, στο, στο σχέδιο γνωμοδότηση, γιατί βλέπουμε να υπάρχουν και περισσότερε επιπτώσει ανάλογα με το φέλλον. Από εκεί και μετά, εμ, εδώ η ε, πρόταση που γίνεται δεν θίγει οι ε, ισχύουσε οδηγίε. Οπότε, καταρχήν, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε ε, θα είναι να ενισχυθούν οι φυστάμενε οδηγίε που ισχύουν για τον κλάδο τη εργασία. Δηλαδή, οι, ε, ε εργαζόμενοι θα πρέπει να εργάζονται μόνο για το χρόνο εργασία για τον οποίο αμείβονται. Γιατί αν εργάζονται για παραπάνω χρόνο, μιλάμε για αθέμητου όρου εργασία, αθέμητε συνθήκε εργασία και αυτό έχει βέβαια με τη σειρά του ανετικέ επιπτώσει στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και προσωπικού βίου. Άρα λοιπόν εδώ το πλαίσιο θα πρέπει να περιλαμβάνει γενικότερα, ευρύτερα κριτήρια, ευρύτερε αρχέ, αν θέλετε, ε, του σωστού, του ορθού και προβλεπόμενου χρόνου εργασία. Από εκεί και μετά, εκείνο που ε, θέλουμε είναι να ληφθεί αυτή η τυχή υπόψη και στο πλαίσιο των κλαδικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των ε, κοινωνικών εταίρων. Κάτι τέτοιο θα πρέπει να τονιστεί ακόμα περισσότερο. Στο άρθρο 18 θα θέλαμε, ή στο σημείο 18 να ε, γίνει λόγος για ε, συχνότερες αξιολογήσεις ε, κινδύνου και να γίνει μια αλλαγή σε ό,τι αφορά την αναφορά και τον υποχρεωτικό χαρακτήρα. Για παράδειγμα, στη δική μου ε, χώρα κάτι τέτοιο είναι υποχρεωτικό μόνο για επιχειρήσει με παραπάνω από 50 εργαζόμενους. Ε, θα μπορούσαμε λοιπόν εδώ ε, να λάβουμε υπόψη μα και τα όσα θα ανακοινωθούν στο πλαίσιο της ε, στρατηγικής ε, τον Ιανουάριο γιατί αυτή τη στιγμή τα όσα προβλέπονται ε, δεν καλύπτουν επαρκώς τις ψυχοκοινωνικές επιτυχίες. Υπάρχουν και ε, κάποια περαιτέρω σημεία τα οποία τώρα δεν θα αναφέρω λεπτομερώς αλλά σε, κάποιες, σε κάθε περίπτωση θα τονίσουμε στις τροπολογίες μας για παράδειγμα το δικαίωμα στην στον ιδιωτικό βίο, ε, την αύξηση της χρήσης, ε, για παράδειγμα, της ε, σύνδεσης στο ίντερνετ και των σχετικών συσκευών, εάν πράγματι ζητείτε από τους εργαζόμενους να είναι πάντοτε συνδεδεμένοι. Και από εκεί και μετά να γνωρίζουμε τι συμβαίνει στις περιπτώσεις εκείνες όπου υπάρχει εξαίρεση από, αυτή την, από αυτό το δικαίωμα για κάποιους εργαζόμενους στην αποσύνδεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει Πρόεδρος, κυρία Σίτλοφ, από το ECR.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 Δεν μεταφράζεται η κυρία Σίτλο. Πρέπει να διακόψω κυρία Σίτλο. okay, okay. Δεν έχουμε εικόνα. Change my camera, okay. Ξέρω, ξέρω. Α, θα πρέπει να αλλάξω θέσεις στην κάμερα. Okay, so we'll continue with uh, the next shadow, the next... Καλώς θα συνεχίσουμε. Ο κύριος Κουσμάου τώρα για την Γκουέντζελ. Και μετά θα επιστρέψουμε και πάλι στην κυρία Τεχόσκη, στην κυρία Τόμ και στην κυρία Σύλλογο. Καταρχήν λοιπόν ο κύριος Κουσμάου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά που έχει κάνει, καθώς έχει συμπεριλάβει πολύ σημαντικά ζητήματα εδώ. Εμείς ε, θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες προκειμένου να ενισχύσουμε μια σειρά από πτυχέ, ε, οι οποίες ήδη αναφέρθηκαν, ή ε, κάποιες από αυτές. Καταρχήν σε ό,τι αφορά τα εργαλεία της τηλεεργασία. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μια καταγραφή αυτών των εργαλείων ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε αυτές τις σχέσεις εργασίας, δηλαδή να μην είναι δυνατό οι εργοδότες να εκμεταλλεύονται με κάποιο τρόπο αυτές τις, ε, αυτές τις συσκευές ε, ψηφιακής εργασίας, τηλεργασίας και επίσης θα πρέπει η συνεργασία και η εργασία που γίνεται από πλευρά των ε, εργαζόμενων να γίνεται ακριβώς μέσω αυτών των εργαλείων προκειμένου να μην υπάρχουν παράλληλες ροές εργασίας. Από εκεί και μετά, επειδή Πρόκειται για έναν τρόπο εργασίας ο οποίος ε, ε, συνεπάγεται ε, ένα μεγάλο βαθμό απομόνωσης των εργαζομένων, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση οι σχετικές οργανώσεις να είναι σε θέση να ορίζουν επακριβώς τους τρόπους ακριβώς τηλεεργασίας. Δηλαδή, θα πρέπει δηλαδή ακόμα και σε περιπτώσει εκείνε που πράγματι χρειάζεται να υπάρχει μια προσαρμογή ε, αυτή των συνθηκών εργασία, θα πρέπει αυτό να συμφορείται και να προβλέπεται επακριβώ. Από εκεί και μετά υποστηρίζουμε πολύ ε, ε, μια ιδέα η οποία ήδη εκφράστηκε ότι δηλαδή το δικαίωμα στην αποσύνδεση θα πρέπει να αποτελεί μια εγγύηση για τους εργοδότες και αυτό σημαίνει ότι για να διασφαλίζεται, για να μπορούμε να εγγυηθούμε πράγματι αυτό το δικαίωμα θα πρέπει να ε, μην είναι δυνατόν να για παράδειγμα να μην προβλέπεται αυτό το δικαίωμα μέσα σε μια συγκεκριμένη σύμβαση εργασίας, αυτό το δικαίωμα στην αποσύνδεση. Δηλαδή σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προβλέπεται. Και από εκεί και μετά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας σε σχέση με το δικαίωμα ε, στην αποσύνδεση ε, και τι των μορφές εργασίας. και το γεγονός ότι δεν θα πρέπει αυτός ο νέος τρόπος εργασίας να αποτελέσει έναν τρόπο με τον οποίο οι εργοδότες θα μεταφέρουν ουσιαστικά το κόστος της εργασίας τους εργαζόμενους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και πάμε στον κύριο Ζεχόφσκι που είναι ο σκιοδησίκτης για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι για αυτήν την έκθεση δεν ξέρω αν πρέπει να συζητήσουμε αυτό το θέμα τώρα, αν είναι τόσο επίγον το θέμα του δικαιώματος αποσύνδεσης, αλλά εντάξει, αυτό συζητάμε τώρα. Έχω κάποια πράγματα να πω για το τι θα θέλει να μπει στην έκθεση αυτή. Καλωσορίζω ότι ανοίγει μια συζήτηση για το θέμα αυτό. Ιδιαίτερα σε αυτή την εποχή όταν η εμπειρία των ανθρώπων που δουλεύουν με τηλεεργασία λόγω της κρίσης, COVID, της κρίσης του COVID είναι πολύ πιο μεγάλη. Είναι όλο και πιο ισχνή η διαχωριστική γραμμή μεταξύ της επαγγελματική και της προσωπικής ζωής και δεν υπάρχει κάποια ευρωπαϊκή νομοθεσία που να καλύπτει το δικαίωμα αποσύνδεσης. Υπάρχουν προσεγγίσεις ε, οι οποίες διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Σε κάποιες χώρες υπάρχουν συγκεκριμένα νομικά πλαίσια, σε κάποιες άλλες ε, υπάρχουν νομοθεσίες που επιτρέπουν την τηλεργασία και υπάρχουν και χώρες που δεν έχουν καθόλου νομοθεσία για το θέμα. Αφενός θέλω να πω ότι βεβαίως και είμαι ότι είναι σημαντικό να υπάρχει αυτό το δικαίωμα αποσύνδεσης και ότι είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα. Είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε την προστασία όλων των εργαζομένων. Από την άλλη, θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε ότι θα λάβουμε υπόψη μας και τις διαφορές που υπάρχουν τις αποκλίσεις από τον έναν τομέα στον άλλον. Σε οικονομικό επίπεδο, σε επίπεδο κλάδου και βεβαίως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, πόσο, εφαρμόσιμο είναι ένα, ένα τέτοιο δικαίωμα. Η υπάρχουσα νομοθεσία θεσπίστηκε σε μια εποχή όπου τα ψηφιακά εργαλεία δεν ήταν και τόσο διαδεδομένα. Οπότε χρειάζεται σίγουρα επικαιροποίηση των κανόνων αυτών. Αυτή η τάση του να είμαστε συνεχώ συνδεδεμένοι, η οποία αυξάνεται, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θα πρέπει να προωθήσουμε αυτό το δικαίωμα αποσύνδεσης και να ζητήσουμε από τις εθνικές αρχές να εισαγάγουν μέτρα, να πάρουν μέτρα που θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό. Θέλω όμως να καταστήσω σαφές ότι δεν είμαι απολύτως πεπισμένος ότι αυτό θα πρέπει να γίνει με κάποιο νέο νομοθέτημα, με κάποιο νέο νομοθετικό μέσο. Τώρα από εκεί και πέρα εγώ είμαι διατηθειμένος να συνεργαστώ με τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε μια πλήρη και σαφή έκθεση. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ζαχώσκη. Και τώρα η κυρία Τάμ από τους Έχετε το λόγο για δύο λεπτά παρακαλώ. Madame Tobe, you have the floor. Παρακαλώ. Sorry, Madam Tom, we can see you, but we... Ναι, σας βλέπουμε, αλλά δεν σας ακούμε, δεν σας ακούμε, κυρία Τόμ. Ίσως να πρέπει να πατήσετε το κουμπί ε, του μικροφόνου. Προσπαθούμε να δούμε γιατί δεν φτάνει ο ήχος στην αίθουσα. Madam Tom, you try Μπορείτε να προσπαθήσετε να μιλήσετε, κυρία Τόμ, να δούμε αν μπορούμε να σας ακούσουμε. Η κυρία Σίμπλε τώρα από την ECR. Κυρία Σίτλερ, έχει το λόγο. Φαίνεται να υπάρχει το ίδιο πρόβλημα. Δεν φτάνει εδώ στην αίθουσα ο ήχος. Μάλλον θα χρειαστεί άλλο ένα πεντάλεπτο διάλειμμα. Προσπαθεί να λύσει το ζήτημα ο τεχνικός. Πέντε λεπτά διάλειμμα. Madame Sander, on va encore une fois tester la connexion parce qu'on a eu un problème avec le son dans la salle. Est-ce que vous voulez euh, presser le... Προσπαθεί γραμματήρια να του με την κυρία Σαντέρ, τη λέει τι να κάνει, μήπω και γίνει η σύνδεση. Voilà. Α, να, λέει η κυρία Σαντέρ. Τώρα με ακούτε καλά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Σα ακούμε πολύ καλά, αλλά και σα βλέπουμε πολύ καλά. Εσεί μα βλέπετε πολύ ωραία. Τέλεια. Οπότε συνεχίστε παρακαλώ. Γεια σα, γεια σα, λέει η γραμματεία. Άρα λοιπόν έχουμε την κυρία Τόμ τώρα η οποία... ωραία. Αυτά με την κυρία Σαντέρ. Ε, περιμένουμε και να δούμε τι θα γίνει με την κυρία Σίντλο. Κυρία Ραφάλσκα επίσης θέλει τον λόγο. Ε, όσο περιμένουμε τους άλλους να σας δώσω τον λόγο. Αλλά ο καθένας από εσάς θα λάβει τον λόγο τώρα. Μιλήστε μόνο ένα λεπτό. Α, η κυρία Τόμ πρώτη. Με ακούτε, ωραία. Συνάδελφοι, ε, και εγώ ε, χαιρετίζω αυτή τη γνωμοδότηση και μου άρεσε η δουλειά που έχει κάνει ο εισηγητής ε, και εγώ θεωρώ ότι από την πλευρά μου κάποιες πλευρές ε, θα χρειαζόμουν να έχω το δικαίωμα και την αποσύνδεση γιατί κάποιες φορές ε, δουλεύουμε το απόγευμα, τα Σαββατοκύριακα και λαμβάνουμε και μηνύματα κατά τη διάρκεια των διακορπών μας και ούτω καθεξής. Οπότε νομίζω πως θα πρέπει να καθορίζεται το δικαίωμα στην αποσύνδεση ε, ανάλογα με και τη φύση της εργασίας. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι κάποιοι άνθρωποι δεν θα έχουν ποτέ αποσύνδεση και θα είναι πάντοτε παγιδευμένοι αν θέλετε με το να έχουν τις συσκευές τους πάντοτε αναμένες. Πάντως θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες. Μετά, σε ό,τι αφορά την ίδια την έννοια της τελεργασίας, να πω ότι και εγώ συμφωνώ με το δικαίωμα που θέλουμε να δώσουμε στους εργαζόμενους να μπορούν να απενεργοποιούν τις συσκευές τους έτσι ώστε μπορούν να, να είναι με την οικογένειά τους ή οτιδήποτε άλλο αλλά αυτό αποτελεί ένα πρώτο βήμα. Δηλαδή, προτού διασφαλίσουμε αυτό το δικαίωμα στην αποσύνδεση, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε καταρχήν το δικαίωμα στη σωστή σύνδεση. Δηλαδή, τι σημαίνει home office. Δηλαδή, όταν έχει κανείς, ε, είναι, βρίσκεται στην οικία του και έχει τρία παιδιά, πώς ακριβώς θα ε, μπορεί να χρησιμοποιήσει την οικία του ως home office. Και μετά, ε, πόσοι άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτόν τον υπολογιστή. Μιλάμε για έναν υπολογιστή, ηλεκτρονικό υπολογιστή που ανήκει στον εργαζόμενο ή του τον παρέχει ο εργοδότης. Ε, ε ο εργοδότης θα πληρώνει, για παράδειγμα, για να έχει ταχύτερη σύνδεση στο ίντερνετ ή ο εργαζόμενος θα κάτι να πληρώσει. Άρα λοιπόν βλέπω ε, πως υπάρχει ε, ο κίνδυνος να δημιουργήσουμε ε, μια νέα φυσιολογική κατάσταση, μια νέα φυσιολογικότητα όπου οι άνθρωποι θα πιέζονται να εργάζονται με αυτόν τον τρόπο όλο ένα και περισσότερο. Ίσως λοιπόν σε ό,τι αφορά ακριβώς αυτήν το, το, το, το είδος της εργασίας του home θα πρέπει να κάνουμε περισσότερες συζητήσεις. Για παράδειγμα, εάν κάποιο έχει για παράδειγμα ε, παιδιά τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται στο σπίτι προκειμένου να ε, ε, φοιτήσουν και εκείνα στο, σχολείο τους διαδικτυακά ένας γονιό θα έχει τη δυνατότητα μόνο να εργάζεται τη νύχτα οπότε πραγματικά αυτό που προσπαθώ να πω με όλα αυτά είναι θα πρέπει καταρχήν να ορίσουμε πιο συγκεκριμένα το τι ακριβώ εννοούμε με την έννοια τηλεργασία και αναμένω με πολύ ενδια... μεγάλο ενδιαφέρον τη συνεργασία που θα έχουμε σχέση με αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ λέει η κυρία Ζήλοφ τώρα από το ECR. Έχει το λόγο παρακαλώ. We'll with... Έχει αποσυνδεθεί η κυρία Σάντερ. Κυρία Σάντερ έχετε μόνο ένα λεπτό στη διάθεσή σα. Και μετά θα δώσουμε το λόγο και στην κυρία Ραφαέλ για ένα λεπτό. Παρακαλώ κυρία Σάντερ. Le droit à la déconnexion est un sujet... Το δικαίωμα για την αποσύνθεση είναι ένα θέμα το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία ακριβώ λόγω τη πανδημία που περνάμε τρώμα γιατί βέβαια η υπόθεση αυτή δεν τελείωσε. Μας περιμένει μια περίοδος ε, αβεβαιότητας ε, σκληρή. Αλλά τέλος πάντων, όποια συνέχεια για να υπάρχει για την πανδημία, νομίζω ότι χρειάζεται ένας νέος τρόπος ε, οργασίας τώρα, ο οποίος θα συνεχιστεί. Και έχουμε και το πολύ σημαντικό θέμα της τηλεεργασίας, οπότε και εμείς θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα θετικά ε, μπορεί να συγκεράσει κανείς περισσότερο επάγγελμα και η οικογένεια. Ε, δεν υπάρχει το στρες της μετακίνησης και λιγότερες εκπομπές διοξιδίου. Ακούγεται πάρα πολύ άσχημα η κυρία Σαντέρ με πολύ ηχό. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να δούμε για την εργασία τι μπορεί να γίνει. Και όλοι θα πρέπει να συνεργαστούμε πάνω σε αυτό, να προβληματιστούμε για το μας στην σε που είναι θεμελιώδες και ακριβώς αποτελεί θεμελιώδες γήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε εγώ θα καταθέσω σχετικά τροπολογίες. Ευχαριστούμε κυρία Σάντερ για αυτό το σύντομο σχόλιο. Κυρία Ραφαέλ Σκατόρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Νομίζω πως αυτό το ζήτημα πραγματικά έχει γίνει πολύ επίκαιρο λόγω της ε, πανδημίας ε, και εγώ συμμερίζομαι τις αμφιβολίες που εξέφρασε μια συνάδελφος. Δηλαδή βρισκόμαστε εδώ στις απαρχές της όλης συζήτηση. Υπάρχουν κάποιες ε, νομοθεσίες σε εθνικό επίπεδο, αλλά γνωρίζουμε ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα θα συνεχίσει να οξύνεται και περισσότερο λόγω της πανδημίας. Εάν λοιπόν προβλέπουμε τις δυνατότητες τηλεργασίας, ε, τότε ενδεχομένως ο, να μπει στον πειρασμό ο εργοδότης να έχει πάντοτε στη διάθεσή του τον εργαζόμενο, αλλά βέβαια ο εργαζόμενος δεν συμφωνεί με κάτι τέτοιο. Βρισκόμαστε δηλαδή ενώπιση ενός διλήμματος αν θέλετε. Γιατί και εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, τόσο και οι βοηθοί μα, όσο και οι εμπειρογνώμονέ μα, όσο και εμεί οι ίδιοι έχουμε πολύ λίγε δυνατότητε να αποσυνδεθούμε. Ε, εξαρτάται λοιπόν το δικαίωμα στην αποσύνδεση και από την καλή οργάνωση της εργασίας. Θα πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε καλύτερα του εργαζόμενου μα ε, και να ευαισθητοποιήσουμε και γενικά κοινή γνώμη σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Γνωρίζουμε πως πολλοί άνθρωποι εργάζονται από τις οικίες τους και αυτό σημαίνει ότι είναι όλο ένα και πιο δύσκολο να έχουν τον απαραίτητο χρόνο για να ξεκουραστούν και είναι ε, ένα και πιο δύσκολο να συμβιβάσουν πλέον τον ιδιωτικό και τον επαγγελματικό βίο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Έχετε πολύ μεγάλο δίκαιο σε αυτό που είπατε ότι δηλαδή και οι βοηθοί μα, το προσωπικό εδώ της γραμματείας, οι εμπειρογνώμονέ μας θα πρέπει να έχουν και εκείνο το δικαίωμα να αποσυνδέονται. Και εμεί το παρέχουμε αυτή τη στιγμή για να είμαστε δικαίοι. Ο κύριος Όλσον τώρα έχει το λόγο. Διευθυντής τη Γενικής Διεθνή Απασχόλησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ, κύριε Όλσον. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο που θίγει αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα και όπως είδαμε στη συζήτηση που έγινε μόλις τώρα πρόκειται για κάτι το πολύ σημαντικό και θα πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω. Ευχαριστούμε επίσης ε, θερμά τον εισηγητή για την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει καθώς θίγει όλες αυτές τις πτυχές. Υπάρχουν ε, μια σειρά από σημαντικά ζητήματα εδώ, γιατί δεν θέλω τώρα να μακρηγορήσω. Υπάρχουν λοιπόν κάποια σημαντικά ζητήματα που και για μας είναι ε, κρίσιμη σημασία. Καταρχήν ο ρόλο των κοινωνικών εταίρων. Οι κοινωνικοί εταίροι θα παίξουν εδώ καθοριστικό ρόλο. Η κυρία ε, Ντεσότερ αναφέρθηκε για παράδειγμα στη συμφωνία πλαίσιο ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ακριβώς κάνει λόγο για αυτή την ε, συμφωνία σε ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση. Αναφέρεται μεν σε αυτήν, αλλά δεν ε, έχει κάποιο κανονιστικό χαρακτήρα. Οπότε θα πρέπει εδώ να λάβουν περαιτέρω δράση οι κοινωνικοί εταίροι. Επίση και οι κλαδικοί κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν περισσότερο σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Και βέβαια, καθώ αυτό το ζήτημα σχετίζεται στενά με την οργάνωση τη εργασία, ε, εμά μα αρέσει πολύ το γεγονό ακριβώ ότι και εδώ η δική σα νομοδότηση θέτει στο επίκεντρο αυτού του ζητήματο του κοινωνικού εταίρου. Κάτι ακόμα πολύ σημαντικό είναι το ότι αυτό που αναφέρεται είναι ότι έχουμε εδώ νομοθεσία, για παράδειγμα, την νομοθεσία σε ό,τι αφορά με το χρόνο εργασία, εκείνο σε ό,τι αφορά τι ε, συνθήκε εργασία που θα ε, τεθεί σε ισχύ του χρόνου και μια σειρά από περαιτέρω ε, νομοθετήματα. Και όλα αυτά θίγουν αυτόν τον τομέα και κατά συνέπεια σε σχέση με οποιαδήποτε πρωτοβουλία θα αναλάβουμε μελλοντικά θα πρέπει να γίνει και σχετική ενημέρωσή του και σωστά αναφέρει αυτό το ζήτημα και ο εισηγητή. και επίσης αναφέρει η κυρία Σάντερ, ναι, το, το ζήτημα τη συζήτηση που θα ξεκινήσει του χρόνου σε σχέση με την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας και ίσως θα είχε νόημα και εκεί να τεθεί. Μετά αναφέρθηκε και το ζήτημα του φίλου από μία σειρά από ομιλητές και εμεί θεωρούμε ότι θεωρούμε πως αυτή η πτυχή θα μπορούσε να αναφερθεί με βελτιωμένο τρόπο μέσα στο κείμενο της γνωμοδότησης και θα μπορούσαμε και εμείς να βοηθήσουμε τον εισηγητή σε ό,τι αφορά περαιτέρω στοιχεία σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Ε, δηλαδή, με βάση και την τελευταία έκθεση που λάβαμε, βλέπουμε πως υπάρχουν μια σειρά από πρωτοβουλίες ε, των ε, κοινωνικών εταίρων, ζητήματα κουλτούρας και των ίδιων των επιχειρήσεων σε έναν ταχαίως μεταβαλλόμενο εργασιακό κόσμο και κατά συνέπεια ακριβώς με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ρυθμιστεί καλύτερα το σχετικό ζήτημα, στο επίπεδο δηλαδή των κοινωνικών εταίρων. Και τέλος έρχομαι ε, στο ε, ζήτημα ε, του ενιαίου αν θέλετε δικαιώματος το οποίο θα ισχύει γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ βλέπουμε μια σειρά από προκλήσει. Προκλήσει σε ό,τι αφορά του κοινωνικού εταίρου, προκλήσει σε ό,τι αφορά την ήδη ισχύουσα νομοθεσία, αλλά και προκλήσει σε ό,τι αφορά τι επιπτώσει στην αγορά εργασία. Δηλαδή, συμμεριζόμαστε εδώ την πρόθεση τη νομοδότηση, αλλά πραγματικά μας προβληματίζει μια τυχόν εφαρμογή του πέραν του πεδίου, αν θέλετε, εφαρμογής των κοινωνικών εταίρων. Ευχαριστώ, λέει η πρόεδρο. Ε, δίνω τώρα το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Σαλίμπα, για να κάνει κάποια καταληκτικά σχόλια. Για δύο λεπτά, παρακαλώ. So, um, first of all, I will... Πρώτα, πρώτα. Ευχαριστώ τους και εισηγητές και όλους τους συναδέλφους που συνέβαλαν. Πολύ θετική και η σημερινή συνεδρίαση. Φάνηκε πόσο σημαντικό είναι το θέμα από τα σχόλια. Είναι πάρα πολύ κακό εγώ του κυρίου Σαλίμπα. Δεν ακούγεται καλά. Θα έχουμε την ευκαιρία τις επόμενες εβδομάδες να μπορέσουμε να βρούμε ένα κοινό παρονομαστή. Να δούμε πώς θα περιχαρακώσουμε αυτό το τόσο θεμελιώδες δικαίωμα. Όπως είπαν όλοι, η πανδημία ανέδειξε περισσότερο μια σειρά θεμάτων. Δεν θέλουμε σήμερα να θεσπίσουμε ένα νέο δικαίωμα. Θέλουμε να ενισχύσουμε υφιστάμενα δικαιώματα που προωθούνται από τους προκατόχους μας, τους συνδικαλιστές μας, δηλαδή το ωράριο εργασίας και άλλα αυτά τα ζητήματα. Τώρα θα πρέπει στεγανά να περιχαργωθούν λόγω της νέας πραγματικότητας. Είναι θέματα που συνδέονται άμεσα και με την ψηφιοποίηση. Θεωρώ ότι το σχέδιο κειμένου μας είναι φιλόδοξο, αλλά από ό,τι διαπίστωσα σήμερα κάποιοι συνάδελφοι σκιώδεις θεωρούν ότι πρέπει να είμαστε πιο τολμηροί Πολύ θετικό αυτό για τη συζήτηση. Και πριν ολοκληρώσω, να σας πω για αυτό που είπε η Πέτρα Ντεσούτερ, που την προβληματίζει. Τα είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώς δηλαδή. Θα προσέξουμε το θέμα της ποιότητας στην έκθεση. Αυτό να περάσει και στο ψήφισμα, αλλά και στην οδηγία ούτως ώστε οι διατάξεις για την ποιότητα να μην μείνουν στην άκρη. Είναι πολύ σημαντικό νομοθέτημα αυτό. Το θέμα είναι πολύ ευρύ. Είναι ένα δικαίωμα που χαρακτηρίζεται από οικουμενικότητα. Αφορά όλους τους εργαζόμενους όλους που χρησιμοποιούν εργαλεία ψηφιακά. Ε, γι' αυτό σας λέω να έχει ευρύ χαρακτήρα και η έκθεση πρόκειται για κάτι για να δικαίωμα πρέπει να απολάβουν όλοι παντού. Τα πράγματα είναι πιο δύσκολα τώρα στην πανδημία αλλά και μετά πιστεύω. Δεν νομίζω ότι θα είναι πεπερασμένη η περίοδος με αυτά τα προβλήματα. Νομίζω ότι και μετά θα υπάρξουν συνέπειες στο μέλλον θα παροξυνθούν τα προβλήματα. Άρα, να είναι ξεκάθαρη με τη ρύθμισή μας η διάκριση μεταξύ χρόνου εργασίας και χρόνου ανάπαυσης. Του χρόνου, όποτε δικαιούται ο εργαζόμενος να απολαύσει την συνέβρεση με την οικογένειά του. Mr. Saliba. The deadline for the amendments 15 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι ε, είναι η ώρα 12 το μεσημέρι είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Περνάμε στο επόμενο σημείο, η θέσπιση μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Ο κύριος Πισλάρου είναι ο συντάκτης αυτής της γνωμοδότησης ε, και δίνουμε λοιπόν τον λόγο στον κύριο Πισλάρου για 8 λεπτά παρακαλώ. Roger, vrei să pleci Hello, can you hear me? Ναι, γεια σας, με ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Ακούμε, αλλά έχουμε και κάτι παράσταση. Uh, now it's better? No, it's some cartoon I'm listening to. Ακούμε Mickey Mouse να παίζει στο background. Α, μισό λεπτό. Can you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 είναι η πραγματικότητα, πρέπει να την πάρουμε και λίγο με χιούμορ. Να αναφερθώ εν συντομία τώρα στο ζήτημα. Στις 28 Μαΐου του 2012 έχει υποβληθεί μια πρόταση για μια, ε, ε, μια, δυνατότητα ανάκαμψης ε, και ανθεκτικότητας. Είναι 90% του προπολογισμού του, του, του Next Generation. Αυτό το το ταμείο, το μέσο έχετε να αντικαταστήσει το προηγούμενο. Το έχουν ξαναζητήσει στην Επιτροπή αυτή. Ο συνεισηγητής αυτού του φακέλου και εγώ παίξα ένα σημαντικό ρόλο για να γίνει αυτή η μετάβαση. Η νέα πρόταση βασίζεται στα τελευταία στοιχεία που έχουμε για μια οικονομική στήριξη των κρατών μελών οι στόχοι έχουν προσαρμοστεί για να λάβουμε υπόψη μας προφανώς τη νέα πραγματικότητα στα πλαίσια του COVID-19 θέλουμε να προωθήσουμε την συνοχή, την οικονομική και την κοινωνική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υπάρξει μια πιο γρήγορη ανάκαμψη με ένα βιώσιμο τρόπο και να είμαστε πιο ανθεκτικοί να μετριάσουμε το κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο της κρίσης του COVID, ταυτόχρονα να υποστηρίξουμε τη μετάβαση προς μια πράσινη οικονομία και την βιώσιμη ανάπτυξη. Πρέπει να έχουμε σχέδια ανθεκτικότητας που να βασίζονται στις προκλήσεις της κάθε χώρας που έχουν εντοπιστεί στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Τα σχέδια αυτά θα είναι επιλέξιμα προς χρηματοδότηση εφόσον συμμορφώνονται με τις ε, συστάσεις του εξαμήνου. Ήθελα να αναφερθώ τώρα στις τροπολογίες που έχουμε υποβάλει και χαίρομαι που θα συμπεριλάβουμε σε αυτήν την ε, αυτό το μέσο και την Χάρτη Θεμελιών δικαιωμάτων, των κοινωνικών δικαιωμάτων. Οι τροπολογίες αυτές θέλουν να υπογραμμίσουν τη σημασία της αλληλεγγύης για την ένταξη, την κοινωνική δικαιοσύνη, την κοινωνική προστασία, αυτό λοιπόν που κάναμε, αφότου είχαμε μια καλή συζήτηση και υπήρξε μια κάποια συνένεση, εγώ επέκτηνα το πεδίο του μέσου στο Άστρο 3 περιλαμβάνοντας μια σειρά από στοιχεία όπως τα μέτρα για την εκπαίδευση, τη διαβίου μάθηση, το καλύτερο, ένα, ένα καλύτερο μέλλον για τα μειονεκτούντα παιδιά, για το τόμα με αναπηρία, ε, αντιμετώπιση της διάκρισης των φύλων, δυνατότητες επιχειρηματικότητας και δημιουργίας δεξιοτήτων, ε, βελτίωση των, των δυνατότητων των δημοσίων αρχών, ε, μέτρα ε, για την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, βελτίωση των συστημάτων υγείας. Μπορέσαμε να συμπεριλάβουμε όλα όσα συζητήθηκαν στις 26 Μαΐου. Έχουμε λοιπόν όλες τις τροπολογίες τις σχετικές που σχετίζονται και με αυτή, αυτό το μέσο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Και βεβαίως αυτό είναι κάτι το οποίο προβλέπεται, δηλαδή αυτή η ενίσχυση για την ανάκαμψη. Οι διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς, με τα εθνικά κοινοβούλια είναι εξελίξη. και βεβαίω υπάρχουν και χώρες ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες αφορά το μέσο. Θα ήθελα να σας ζητήσω να έχετε κατά νου όταν θα υποβάλλετε τις τροπολογίες σας ότι έχουμε κάνει μια πλήρη δουλειά για να, να επεκτείνουμε, να διαβρύνουμε το πεδίο αυτού του μέσου Ιδιαίτερα τα άρθρα 3 και 4 μιλάνε πλέον για έξι πυλώνες. Μετά από μια χαρτογράφηση του τι συμβαίνει στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, έχουμε τους έξι πυλώνες, πράσινη ε, μετάβαση, θεσμική αθεκτικότητα και δύο πυλώνες που έχουν πολύ μεγάλη σημασία να ξεπεράσουμε τις κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας και να υποστηρίξουμε την κοινωνική συνοχή, ο πυλώνας κοινωνικής συνοχής, βασίζεται στην ε, χάρτα κοινωνικών δικαιωμάτων και βεβαίω ο πυλώνα τη νέα γενιά του Next Generation. Βλέπετε λοιπόν ότι η πρόθεσή μας από την αρχή ήταν να τα συμπεριλάβουμε όλα αυτά στην τελική έκθεση. Είμαι στη διάθεσή σα για, για οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε για αυτό το πολύ σημαντικό φάκελο. Αναμένουμε ανυπομονησία να συνεργαστούμε εκ νέου για το φάκελο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Ντράγκος. Και τώρα να περάσουμε στους κοιόδης συζητητές. Δύο λεπτά ο καθένας παρακαλώ. Ξεκινούμε με το ΕΛΚ. Ο κύριος Φερνάντες έχει το λόγο. Στα πορτοκαλικά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή ε, με τον οποίο είχα τη δυνατότητα να εργαστώ σε αυτό το τομέα σε σχέση με, αυτήν την, ε, ε, με αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. Ε, είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό το ταμείο του Μηχανισμού Ανακαμψής και Ανθεκτικότητας να εγκριθεί το ταχύτερο δυνατό. Και για να γίνει αυτό θα χρειαστεί λοιπόν καταρχήν να εγκριθεί ο σχετικός μηχανισμός. Ελπίζουμε οι σχετικέ διαδικασίε στα εθνικά κοινοβούλια, δηλαδή η κύρωση και οι ίδιοι πόροι να είναι δυνατό να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατό για να ξεκινήσει και η κροή των σχετικών κοντιλίων το ταχύτερο δυνατόν. Θέλουμε μια Ευρώπη συνεργατική, ανθεκτική και για να το επιτύχουμε αυτό θα πρέπει οι μικρομεσαίε επιχειρήσει, οι οποίε είναι και εκείνες που δημιουργούν ε, τελικά τις περισσότερες θέσει εργασία, να λάβουν την κατάλληλη υποστήριξη. Επίση, θα πρέπει να ενισχύσουμε την οικονομική, κοινωνική και εδαφική σύνοχη τη Ευρω... Ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις ε, σχετικές τροπολογίες που έχω υποβάλει 21, 22, 23, είναι εξαιρετικά σημαντικό να δώσουμε έμφαση στην επιχειρηματικότητα. Κάτι ακόμα που θα ήθελα να αναφέρω είναι ένα εργαλείο τεχνικής υποστήριξης το οποίο σχετίζεται με αυτό το, το μηχανισμό ανάκαψης και ανθεκτικότητας. Οπότε δεν θεωρώ εγώ πως αυτό το, τα κονδύλια τα οποία προορίζονται για αυτόν τον μηχανισμό να κατευθυνθούν για παράδειγμα για την υποστήριξη σεμιναρίων τη χρηματοδοτική. Όχι, για κάτι τέτοιο έχουμε το, ακριβώς το τεχνικό εκείνο εργαλείο το σχετικό κονδύλιο. Και από εκεί και μετά, εάν τα κονδύλια ε, που προβλέπονται για ε, το μηχανισμό ανάκαψης και ανθεκτικότητας δεν απορροφηθούν, τότε θα μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν για να μην χαθούν σε προγράμματα τα οποία ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου υπάρχει δηλαδή τεράστια προστιθέμενη αξία, για παράδειγμα στο ε, Erasmus ε, Plus, ε, στο Horizon 2020 και ούτω καθεξή. Δεν ξέρουμε κατά πόσο δηλαδή, τα κράτη-μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να απορροφήσουν όλα τα κονδύλια όπω αυτά προβλέπεται στο μηχανισμό ανάκαμψη και ανθεκτικότητας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε σε θέση να επαναχρησιμοποιήσουμε, να επαναξιοποιήσουμε τα σχετικά κονδύλια για ευρωπαϊκά προγράμματα όπως ε, ανέφερα το Erasmus Plus για παράδειγμα, το Horizon 2020 ή και το Invest EU, το οποίο έχει και δεχθεί μια μεγάλη περικοπή. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να εστιάσουμε λίγο παραπάνω στον τομέα της εφαρμογής ε, στην πράξη αυτού του μηχανισμού και αυτό θα πρέπει να αναφερθεί και περισσότερο στο σχέδιο γνωμοδότηση σε σχέση με τις προτάσεις που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και στην α, τοπολογία 35 εκεί ε, γίνονται κάποιες ε, προτάσεις ε, σε ό,τι αφορά την επιστροφή κάποιων κονδυλίων στα κρατημέρια, γιατί δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό θα είναι δυνατόν να απορροφηθούν και να αξιοποιηθούν με τον σωστό τρόπο όλα αυτά τα κονδύλια μέσα σε βάθος τριών ετών. Yes, thank you. Thank you. Κυρία Ντόμπρε, ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτό το μέσο ανά, ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο των, του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μέσω των συστάσεων ανά χώρα. Το να συνδέσουμε το μέσο με το εξάμεινο θα δώσει κίνητρο στα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν ε, τις ελλείψεις που αντιμετωπίζουν. Ε, αυτή τη στιγμή τα κράτη-μέλη έως τώρα ήταν αρκετά ε, διστακτικά στον εφαρμόσουν τι συστάσει αναχώρα και ίσω αυτό να αλλάξει τώρα. Κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά, σημαντικό εδώ είναι ότι αν ένα κράτο μέλο δεν κάνει επαρκεί προσπάθειε, ε, τότε μπορεί η χρηματοδότηση να διακοπεί. Και αυτό μπορεί να εξασφαλίσει τελικά ότι θα λάβουν χώρα αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Είχαμε ε, σημαντικές ελλείψεις στην πρόταση της Κομισιόν, ε, παραδείγματος χάρη ε, ότι πέρα από την πράσινη και την ε, ψηφιακή μετάβαση δεν υπήρχε κοινωνική διάσταση. Έλειπε παντελώ. Δεν υπάρχει καμία καθόλου αναφορά στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Πώ θέλουμε μια ανθεκτική οικονομία χωρί μια ισχυρή ε, κοινωνία, ιδιαίτερα μετά την ε, κρίση του COVID. Χάρηκα λοιπόν που είδα το έργο του εισηγητή και χάρηκα ιδιαίτερα με την προσέγγιση του. Νομίζω ότι έχουμε κάνει μια καλή δουλειά ε, το Μάρτιο ή το Μάιο καλύτερα ε, σε ό,τι αφορά το σχέδιο υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων ε, δύο, χρόνια, δύο μέρες μάλλον μετά την, την εκπόνησή του προχώρησε στην Ομόδια Επιτροπή έχει βελτιώσει σημαντικά ο εισηγητής στο αρχικό κείμενο έχει συμπεριλάβει κοινωνικούς δείκτες που συνδέουν τους στόχους του μέσου με τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και νομίζω, και νομίζω ότι για όλους μας είναι σημαντικό να υπάρχει μια πιο ευρία συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα κράτη-μέλη τα οποία πρέπει να έρθουν σε επαφή με τους κοινωνικούς εταίρους πριν ε, σχεδιάσουν το σχέδιο ανάκτησης και ανθεκτικότητας, δεν μπορεί να υπάρξει ανάκαμψη χωρίς ισχυρό κοινωνικό παράγοντα. Εγώ χαιρόμαι ιδιαίτερα προσωπικά ότι το κείμενο αυτό ε, προβλέπει διακοπή ε, όταν ένα κράτος μέλος δεν συμμορφώνεται. Ε, ιδιαίτερα ε, όταν υπάρχουν και προβλήματα με το κράτος δικαίου σε κάποιες χώρες. Θα υποστηρίξω λοιπόν αυτές τις τροπολογίες, ε, θα υποβάλουμε και κάποιες να συμπεριλάβουμε τη δημιουργία των κοινωνικών εταίρων, διότι δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν ε, ε δεν υπάρχει ισχυρή εταιρική σχέση των κοινωνικών εταίρων αν δεν υπάρχουν ισχυροί κοινωνικοί εταίροι. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ντάμπρεκ και τώρα συνεχίζουμε με την ID. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Αγγέλα Μέρκελ ε, υποσχέθηκε ότι όσο θα ζει δεν θα υπάρξουν χρέη σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. αλλά φαίνεται να είπε για μία ακόμα φορά ψέματα στον ε, ε, στο λαό της. Ε, δηλαδή, ο Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας ε, είναι πιο ειλικρινής και είπε ότι μπορούμε να έχουμε περισσότερα χρέη και όλο και περισσότερα χρέη και τώρα αναφερόμαστε και σε ίδιους πόρους, για παράδειγμα, μέσω του συστήματος εμπορίας εκπομπών. Αλλά όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν με τις συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν σχετίζονται με αυτά και ούτε προβλέπονται στις συνθήκες ούτε και στην νομοθεσία. Αλλά από ό,τι φαίνεται κανεί δεν ενδιαφέρεται για όλα αυτά. Εμεί τελικά διαμορφώνουμε τα πράγματα έτσι όπω μα αρέσει. Φυσικά και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της πανδημίας. Αλλά αυτό το, αυτός ο μηχανισμός ε, ανάκαμψης ε, είναι ουσιαστικά ε, πεταμένα λεφτά. Και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει και ο γνωστός οικονομολόγος Γιώργεν Μάρτης. Γιατί ποιος τελικά θα υποφεληθεί περισσότερο από αυτά τα κοντήλια, η Ελλάδα και η Βουλγαρία. Και δεν νομίζω ότι η Ελλάδα και η Βουλγαρία έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την πανδημία. Τουλάχιστον δεν έχω αυτή την αίσθηση. Άρα λοιπόν εγώ νομίζω πως πλέον βρισκόμαστε στη φάση ολοκλήρωσης ε, της Ένωσης ε, Χρεών. Και εμεί δεν θέλουμε να συμμετάσχουμε σε αυτό. Ε, ο οικονομολόγο κ. Ζήμ και καθηγητή αναφέρει το ότι το 16% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωση δεν βρίσκεται πλέον σε, σε συνθήκες ζωής κατάλληλες. Αλλά κάτι τέτοιο είναι πρωτόγνωρο. Δεν μπορούμε να, να επιβιώσουμε αυτόν τον τρόπο σε ένωση. Άρα λοιπόν σε ορισμένε περιπτώσει βλέπουμε κάποιοι να καλούνται μόνο να πληρώνουν και να μην λαμβάνουν καμία υποστήριξη από την Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Πίτερ Χάνσεν για τους πράσινους. Can, now you can see and hear me, right? Yes, we can hear you, we can see you. Yes, okay. Ναι, ναι, και σας βλέπουμε και σας ακούμε. Ευχαριστούμε τον εισηγητή και τους όλους αδέλφους, τον κύριο Πισλάρο. Έγγελα Μέρκελ και άλλοι πολιτικοί ανέλαβαν τις ευθύνες τους. Άκουσα τι είπε ο συνάδελφος από το έδικ και θα πρέπει να το πω αυτό. Θα πρέπει κάτι να γίνει για τις επιπτώσεις του κορονοϊού. Και υπάρχει πρόβλημα στις, στις ε, επιχειρήσεις, στην οικονομία. Γι' αυτό και είναι σημαντικό το ότι θεσπίστηκε ε, αυτός ο μηχανισμός ανακαμψής και ανθεκτικότητας. Νομίζω θα υπάρξουν συνέπειες για την ευρωπαϊκή οικονομία, να σταθούν ξανά στα πόδια επιχειρήσει και έτσι επίση να δοθεί μια ευκαιρία στι μέλουσε γενιέ. Οπότε γι' αυτό, ε, για να το εξασφαλίσουμε, θα πρέπει το μηχανισμό αυτό να είναι ουδέτερο, από πλευρά ε, διοξιδίου, να ευθυγραμμιστεί με το New Green Deal, άρα χρειαζόμαστε ε, όσον αφορά τον μηχανισμό ε, δεσμευτικούς στόχους και να είναι ανάλογες και να που θα γίνουν στα πλαίσια του μηχανισμού. Άρα να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει δημοκρατικός έλεγχος και ότι θα ισχύσει το κράτος του δικαίου. Και άρα να έχουν πρόβλημα τα κράτη τα οποία δεν σέβονται τις δημοκρατικές αξίες. Να μην καλυφθούν. Βεβαίω στα πλαίσια αυτά να ληφθεί υπόψη ισότητα ανδρών γυναικών. Μπράβο που διεύρυνε ε, το κείμενο ο εισηγητής. Λοιπόν, να περιμένω τη συνέχεια των εργασιών μας και ελπίζω ότι θα συμβιβαστούμε, θα βρούμε κοινό παρανομαστή για μέρους ζητήματα ε, και έτσι θα εκπροσωπήσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες από κοινό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πίτερ Χάνσεν και τώρα η κυρία Ραφάλσκα για το ECR. Ευχαριστώ. Λέει η κυρία Ραφάλκα. Ευχαριστώ και τον κύριο Πισλάρου που και πάλι έχει προετοιμάσει ένα κείμενο πλήρες. Μπορεί να πει κανείς ότι διατηρεί αμφιβολίες για αυτό τον μηχανισμό. Είναι τέλειος. Έτσι θα ενισχυθεί η ευρωπαϊκή οικονομία και η ανθεκτικότητα γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, με δεδομένη την παρουσία της πανδημίας είναι ακόμα πιο σημαντικός αυτός ο μηχανισμός. Έτσι θα υποστηριχθούν και οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις. Όπως τα πράγματα είχαν πριν, χωρίς δηλαδή τέτοιους μηχανισμούς, οι χώρες εκτός Ευρωζώνης δεν είχαν βοήθεια για επενδύσεις, για την Ήπεθρο, για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές τους. Ε, για αυτό και ήταν μειωμένη η δυνατότητα για επενδύσεις. Αν δεν αναφέρεται της ανθεκτικότητας ε, των περιφερειών και ο εισηγητής. Επίση μα μιλά και για αυτό το εργαλείο, αυτό το μέσο τεχνική αρρωγή. Πάντω, θα πρέπει να μην είναι πολύ περιοριστικοί οι κανόνες, οι διατάξεις ε, αυτού του μηχανισμού, γιατί έτσι θα περιοριστεί και η υποστήριξη για κάποιους τομείς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Ε, η κρίση της ε, πανδημίας ε, κατέδειξε κάποιες από τα, κάποτα ευαίσθητα σημεία, τα ευάλωτα σημεία στην Ένωση και νομίζω πως αυτός ο μηχανισμός μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει εκείνο που είχε προβλεφθεί και το οποίο κάνει συγκεκριμένες ε, προτάσεις ε, χωρίς όμως να έχουμε καταφέρει να φτάσουμε ε, σε μια δυναμική οικονομική ανάπτυξη και δεν καταφέραμε να αναστρέψουμε την μείωση των θέσεων εργασίας. Δεν θέλουμε λοιπόν μια πολιτική η οποία είναι απορριθμιστική και εφαλοκρατική και η οποία τελικά μειώνει τα δικαιώματα των εργαζόμενων. ξέρουμε ποιε είναι οι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει και ποιο είναι ο αρνητικό αντίκτυπο που έχουν στι ζωέ των πολιτών. Αυτό λοιπόν που χρειαζόμαστε είναι πολιτικέ οι οποίε υπερασπίζονται του μισθού και τα δικαιώματα εργασία των εργαζόμενων ε, και επίση υποστηρίζουν τη συνέχιση τη παροχή δημόσιων υπηρεσιών ε, για όλου ε, και δωρεάν θα πρέπει να έχουμε σωστά μέτρα για να έχουμε την κατάλληλη λήψη μέτρων προκειμένου να αποφύγουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ε, και οι τροπολογίες που εμείς θα ε, υποβάλλουμε θα κινηθούν ακριβώς σε αυτόν τον άξονα. Ευχαριστώ. Έχουμε μαζί μας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και την κυρία Ντρές. Θέλω να της δώσω ευθύς αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Συγητή, αξιότιμα μέλη, θέλω να σε ευχαριστήσω που μας δίνετε το λόγο για να συνεισφέρουμε και εμείς εν συντομία σε αυτή τη συζήτηση. Θα θέλαμε να σας δώσουμε μια πρώτη αντίδραση μετά τις παρεμβάσεις των ομιλητών και το σχέδιο γνωμοδότησης του Συγητή, Τον ευχαριστούμε για αυτό. Αναγνωρίζει ε, ότι η πρόταση αυτή μπορεί να συνεισφέρει σε μια ανάκαμψη όσο γίνεται πιο γρήγορα. Θέλουμε να προχωρήσει γρήγορα και το κείμενο βέβαια. Σε ό,τι αφορά τον στόχο και τον σκοπό θα συνεισφέρει στην εφαρμογή του κοινωνικού πυλώνα βεβαίως αυτή η προσπάθεια ε, λόγω των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 4 για τον κοινωνικό τομέα και βεβαίως θέλουμε να προωθήσουμε την οικονομική, κοινωνική και εδαφική ε, συνοχή και να μετριαστούν τα αποτελέσματα της κρίσης. Ξέρουμε ότι το ERF δεν εξετάζει μόνο την ανάκαμψη, εξετάζει και το μέλλον, μιας και θα χρειαστούν μεταρρυθμίσεις στα πλαίσια του Next Generation ε, και βεβαίως υπάρχει η ψηφιακή μετάβαση και η αύξηση της ανθεκτικότητας. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτά που αναφέρει ο συγκητή στι τροπολογίε του, όπω η βελτίωση των δεξιοτήτων, η προσέγγιση των επιχειρηματιών, ήδη καλύπτονται από τον κανονισμό ω έχει. Έτσι λοιπόν, θέλουμε να ενθαρρύνουμε την Επιτροπή σα να μην προσθεθούν πολλά πράγματα σε επίπεδο στόχων, διότι αυτό θα είναι αντιπαραγωγικό. Θα νερώσουν το μήνυμα. Το πεδίο ως έχει ε, τώρα είναι επαρκέ, είναι σαφέ και θα οδηγήσει σε επενδύσεις ε, για ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά για αυτή την Επιτροπή. Ε, λαμβάνουμε γνώση ε, της, σημασίας που θέλει να δώσει η Επιτροπή στην ε, διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, μεταξύ των οποίων κοινωνικού εταίρους. Θέλουμε βεβαίως να υπάρξει μια προτεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που αναφέρονται και βεβαίω χρειάζεται διαβούλευση με τι εμπλεκόμενου φορεί για να συμβεί αυτό. Δεν μπορούμε να παρέμβουμε στι εθνικέ διαδικασίε βέβαια, μπορούμε όμω να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να προβούν σε αυτέ τι διαβουλεύσει, χωρί να χρειαστεί παρόλα αυτά να αλλάξει η νομοθεσία. Θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι έτσι όπω αντιλαμβανόμαστε εμεί τη φύση των αποφάσεων που θα πρέπει να πάρθουν στα πλαίσια του ERF, ε, το κατάλληλο νομοθετικό μέσο είναι μια ε, ε, καταξιδότηση πράξη είναι κάτι το οποίο θα αναφέρει τα διάφορα στοιχεία της νομοθεσίας, θα τα διευκρινίσει ε, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας, χωρίς να προσθέτουμε νέους κανόνες και χωρίς να ε, επηρεάζεται και να αλλοιώνεται ουσιαστικά το κείμενο. Δεν πρέπει να επιβαρύνουμε υπερβολικά το κείμενο. Οι εκθέσεις προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο προβλέπονται ήδη στην πρόταση, η αναφορά προς τα όργανα αυτά. Επίσης θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή της Επιτροπής σας ότι οι επενδύσεις ε, πάνε χέρι-χέρι με την προσπάθεια αυτή που γίνεται. Οι κοινωνικές επενδύσεις θα είναι κλειδί για τους κοινωνικούς στόχους ε, ε, που έχει θέσει το μέσο. Σας ευχαριστώ πολύ για την δέσμευσή σας γύρω από αυτό το φάκελο. Ευχαριστώ πολύ και τώρα το λόγο έχει εκ νέου ο εισηγητής για τα για τελευταία σχόλια. Κύριε Πισλάρο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, όντως έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία. Να πω δύο-τρία πράγματα σε σχέση με αυτά που αναφέρθηκαν. Συμφωνώ πολύ με τον συνάδελφο τον κύριο Φερνάντες από το ΕΛΚ. Θα πρέπει να κινηθούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και συμφωνώ απολύτω ότι η επιχειρηματικότητα, η κοινωνική επιχειρηματικότητα, οι μικρομεσαίε επιχειρήσεις είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο ε, και εμεί το υπογραμμίσαμε αυτό. Σε ό,τι αφορά αυτό που είπε ο κ. Καραντόφ, χαίρομαι που μπορέσαμε να προωθήσουμε κάποια από τα στοιχεία αυτά και εμείς θέλουμε η δημιουργία δυνατοτήτων να είναι επιλέξιμη στα πλαίσια της θεσμικής ανθεκτικότητας και του σχετικό πυλώνα και αναμένω και τις υπόλοιπες τροπολογίες που μας προαναγγείλατε. Σε ό,τι αφορά αυτά που είπε ο Πίτερ Χάνσεν από τις Πράσινους, Συμφωνώ απολύτως ότι είναι μια ευκαιρία αυτή που εμφανίζεται μια φορά μόνο. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την ε, ισότητα των δύο φύλων, την εκπροσώπηση των δύο φύλων και βεβαίως θα πρέπει οι αρχές μας ε, να είναι σαφείς για τα ζητήματα αυτά στο κείμενο. Σε ό,τι φορά την παρέμβαση την κυρία Φραντσέσκα από το ECR είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα ε, πεδίο ανταγωνιστικότητας ισότιμο για όλους και βεβαίως πρέπει να δώσουμε τεχνική υποστήριξη προς τα κράτη-μέλη εκείνα που την χρειάζονται. Σε ό,τι αφορά την παρέμβαση της κυρία Περέιρα από την ΚΟΕ, έχουμε υπογραμμίσει σαφώς και πολύ συγκεκριμένα ότι η κοινωνική ε, και η διαρθρωτική Εντάξει, είναι πολύ σημαντική. Ξέρουμε ότι η αλληλεγγύη αυξάνει την ανθεκτικότητα και τη δυνατότητα που έχει μια κοινωνία να αντιδράσει απέναντι σε τέτοια σοκ. Ευχαριστούμε την Κομισιόν για τη συμμετοχή και την αντίδραση. Συμφωνούμε με πολλά από αυτά που είπατε. Χαίρομαι που θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε και βεβαίως έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα κάνει μια εφαρμογή προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που θέλω να υπογραμμίσω σε σχέση με την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όμως. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι εμείς δεν θέλουμε απαραίτητα μια πράξη κατεξιοδότηση επειδή δεν, δεν ε, εμπιστευόμαστε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρόβλημα είναι ότι το Συμβούλιο το καλοκαίρι πήγε προς μια διακυβερνητική προσέγγιση όπου τα κράτη-μέλη θα έχουν λόγο για, για πολύ συγκεκριμένα ζητήματα ε, που κανονικά θα πρέπει να αποφασίζονται σε επίπεδο κομισιών. Μια και υπάρχει αρχή τη συναπόφαση και επειδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ε, αυτή, το, αυτό το δικαίωμα στην απόφαση με το Συμβούλιο, είναι πολύ σαφέ για μα ότι το Συμβούλιο είναι αυτό το οποίο θα ασχοληθεί με την ουσία και εμείς απλώς θα κάνουμε κάποιες ακροάσεις. Θα υπογραμμίσουμε λοιπόν ε, το, τη σημασία του ρόλου του Κοινοβουλίου εδώ, διότι εμείς εκπροσωπούμε τους πολίτες, είμαστε εκλεγμένοι, είναι πολύ σημαντικό αυτό για να μειωθεί και το δημοκρατικό έλλειμμα. Δεν είναι θέμα εμπιστοσύνη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς εμπιστευόμαστε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε την, ορ, την ορθή βάση διακυβέρνησης. Ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογής, ε, είναι η βασική ε, αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο σχεδιασμό του μέσου αυτού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό ε, για μα. Ελπίζουμε η Κομισιόν να κάνει καλή δουλειά και την εμπιστευόμαστε στην εφαρμογή. Όμω, προ όφελο των συμπολιτών μα, πρέπει στο πεδίο και στου στόχου να υπάρχουν κατευθυντικέ γραμμέ οι απαραίτητε, έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρξει πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Και θα έχουμε τι σωστέ προτεραιότητε, έτσι ώστε να έχουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση, μια σωστή απάντηση απέναντι στην πανδημία και οποιαδήποτε άλλα σοκ μα περιμένουν στο μέλλον. Θεωρούμε ότι γι' αυτό δίνουμε έμφαση στην ανάκαμψη και στην ε, ανθεκτικότητα για τους πολίτες μας. Σας ευχαριστώ πολύ για το έργο που κάνετε, που κάνουμε όλοι μαζί. Η Επιτροπή ΕΜΠΛ θα συνεισφέρει, πιστεύω, κατά πολύτιμο τρόπο στην ε, ολοκλήρωση του φακέλου αυτού. Σας ευχαριστώ πολύ για την ολοκλήρωση του θέματος αυτού. Να σας θυμίσω ότι 10 Σεπτεμβρίου είναι η προθεσμία για τι τροπολογίε. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη, που είναι και το τελευταίο. Είναι το σχέδιο γνωμοδότηση ε, για τι νέε οδού νόμιμη μετανάστευση. Η κυρία Ραφάλσκα είναι η συγγήτρια από το ECR, ε, την οποία θα ακούσουμε ευθύ αμέσω. Θα μα παρουσιάσει το σχέδιο έκθεση. Κυρία Ραφάλσκα, έχετε 8 λεπτά στη διάθεσή σα, παρακαλώ. nowe drogi legalnej migracji pracowników. E, η κυρία Ραφάλσκα. Μιλούμε τώρα για νόμιμη μετανάστευση για λόγου εργασία. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δούμε πώ θα υπάρξουν νέοι διάβλοι. Ε, μεγάλο το πρόβλημα, αλλά δύσκολη και αυτή η έκθεση. Δεν πρόκειται για ένα νέο φαινόμενο. Αυτά ε, είναι θέματα των Τα μάρτυρε εδώ και δεκαετίε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οπωσδήποτε μια που ε, προχωράει η τεχνολογία και οι τηλεπικοινωνίες ε, ε, εντείνεται αυτό το φαινόμενο οπότε και είναι και ακόμα πιο ε, σημαντικό για τις εθνικές αγορές εργασίας δεν έχουμε στατιστικές που να δίνουν την πλήρη εικόνα για την μετανάστευση και αναφέρεται ότι την περίοδο 9 έως 19 είχαμε 19 με 20 εκατομμύρια νομίμων μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να, έτσι βλέπετε ε, την κλίμακα, το μέγεθος του προβλήματος και ακόμα και αν είχαμε την ε, αρμοδιότητα για να θεσπίσουμε τους όρους και προϋποθέσεις ε, εισόδου των ηθαγενών τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό αφορά την επανένωση οικογενειών. Και βέβαια τα κράτη-μέλη διατηρούν το δικαίωμα να αποφασίσουν όσον αφορά ε, τον όγκο της μεταναστευτικής ροής. Για αυτούς δηλαδή που αναζητούν εργασία στην επικρατεία τους, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, να ε, υιοθετούν μια προσέγγιση που έχει σχέση με ε, αναλύσεις, ποσοστώσεις και έτσι καθορίζουν λοιπόν τα σχετικά κριτήρια. Καλό να έχουν τέτοια αυτονομία τα κρατημέλη, είναι μεγάλο το πρόβλημα και είναι αδύνατο να καλυφθούν όλα τα θέματα ε, σε μια τέτοια πρώτη γνωμοδότηση. Έχουμε επίσης τα σχετικά με το περιορισμό για την έκταση της έκθεσης. Τέλος πάντων, ελπίζω ότι όλα θα ξεκαθαριστούν και ελπίζω να συνεργαστώ με τους σκιώδους ηγητές και να είναι αξιόλογο το κείμενο για την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Τώρα όσον αφορά το θέμα των δημογραφικών προβλημάτων. Ε, αυτή την επιτυχία του Δήματος έπρεπε να την καλύψω, διότι όταν μιλούμε για αγορά εργασία και για τα σχετικά προβλήματα, θα πρέπει να μην ξεχνούμε και τα δημογραφικά. Ότι δηλαδή είναι γυράσκωσες οι κοινωνίες μας, ότι υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού. Να τα βασικά προβλήματα για πολλούς κλάδους. Αυτοκινητομηχανίες, ε, οικοδομή κλπ. Όλα αυτά αλληλό συνδέονται. Υπάρχει αλληλεξάρτηση. Επίσης, από την μεριά, η Ευρωπαϊκή Ένωση ελκύει εργαζόμενους με λιγότερες δεξιότητες από όσο θα ήθελε, από όσο θα περίμενε. Οπότε αυτό τώρα είναι θέμα για τα κρατημέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να διαφημίσουν αγροεργασία ω μια εργασία ενδιαφέρουσα και ελκυστική. Θα πρέπει επίση να προωθήσουν ε, τι θέσει μα. Η μετανάστευση είναι απάντηση στα σημερινά προβλήματα, άπαξ και οι μετανάστες είναι στη θέση να εργαστούν στους τομεί για του οποίου έχουν δεξιότητες. Εγώ είμαι Πολωνέζα και πάρα πολλοί συμπατριώτες μου φύγαν από τη χώρα γιατί αναζητούσαν καλύτερη δουλειά στο εξωτερικό. Και επίσης αναζητούσαν και καλύτερη αμοιβή. συνήθω εκτιμώνται γιατί είναι φιλότιμοι, δουλεύουν σκληρά και πολλοί από αυτούς έχουν όμως ε, πάρει δουλειές και κάνουν δουλειέ που δεν αποκρίνονται στι δεξιότητε, στα προσόντα του. Κυρίω αυτό ή στο παρελθόν. Ε, γι' αυτό σα λέω ότι έτσι δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το ανθρώπινο κεφάλαιο. Πάει χαμένη η παιδεία, η εκπαίδευσή τους, οι οξιότητές τους. Επίσης έχουμε και ένα φαινόμενο φυγής εγκεφάλων, γιατί πάρα πολλοί με προσόντα εγκαταλείπουν τη χώρα τους. Και Βέβαια, αυτό έχει σχέση με το τι κατάσταση επικρατεί στην αγορά εργασίας της χώρας του καθενός. Οπότε, μπορεί σε κάποια χώρα ήδη να υπάρχει μεγάλη ενεργεία ή μπορεί να υπάρχει πλήρης αποσχόληση και μπορούν να υπαγορεύσουν τις συνθήκες που θέλουν οι εργοδότες. Τώρα στον καιρό τη επιδημία αναδείχαν πολλά προβλήματα που προπήρχαν, όπως πούμε η ελευθερία της παροχής υπηρεσιών. Τα έχουμε συζητήσει αυτά στην Επιτροπή. Όταν συζητούσαμε για τους εποχιακούς, το πρόβλημα παραμένει. είναι το θέμα της ε, διαμονής τους ε, σε μια χώρα αυτών των ε, εποχιακών ή τον ασχολούμενο με την πληροφορική και θα πρέπει να δούμε τι πρότυπα υπάρχουν για την κινητικότητά τους και για το πρόβλημα του ότι πολλές φορές έχουν βιωτικές συνθήκες πάρα πολύ άσχημες αυτοί οι εργαζόμενοι. Άλλο σημαντικό είναι η καταπολέμηση του του ανταγωνισμού. Γιατί εδώ στην Επιτροπή μας ασχολούμαστε με τον κοινωνικό πυλώνα και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η δουλειά είναι μια αφετηρία. Ότι ε, ε, αν έχουμε μια καλή δουλειά τότε μπορούμε εκεί να υλοποιήσουμε αυτά τα οποία έχουμε μάθει και μπορούμε να, έτσι να καταπολεμήσουμε ε, της δυσμενής διακρίσης, να μην υπάρχει στιγματισμός, ε, γιατί αλλιώς ε, έτσι οδηγούμαστε σε διάπραξη εγκλημάτων. Το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό σας λέω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια καλή συνεργασία με τους κοιόδης συζητητές και νομίζω ότι ειδικά το θέμα αυτό έχει μέλλον μπροστά του. Γι' αυτό σας λέω, ελπίζω να είμαστε θετικοί και όποιος θέλει να υποβάλει τροπολογίες, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου μπορεί να μας ε, τις υποβάλει η Πρόεδρος τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εισαγωγή που κάνατε, κυρία Πραφάλσκα. Και τώρα το λόγο έχουν οι σκιώδες και πρώτος πρώτος ο κύριος Κάνεφ για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. can we hear each other well? Yes, we can. Καλημέρα, μας ακούτε? Με ακούτε καλά, ωραία. Ε, σας χαιρετώ από τη Σόφια και ευχαριστούμε ε, εδώ την εισηγήτρια την κυρία Ραφάλσκα για αυτό το πρώτο σχέδιο νομοδότησης. Ε, θα πω πολύ λίγα πράγματα έτσι ώστε να υπάρχει περισσότερος χρόνος για τη συζήτηση που θα κάνουμε. Να πω ότι πρόκειται για μια πολύ καλή βάση για περαιτέρω συζήτηση έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια καλή γνωμοδότηση της ΕΜΠΛΕ για αυτό το ζήτημα. Και για μένα δύο τεινά είναι τα πιο σημαντικά και προς αυτή την κατεύθυνση προετοιμάζω τις τροπολογίες μου και αυτά είναι τα εξή. Χρειαζόμαστε μία πιο ξεκάθαρη και άμεση προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι να έχουμε περισσότερη και καλύτερη εντοενωσιακή κινητικότητα των εργαζόμενων βλέπουμε ότι αντιμετωπίζουμε κυρίως το ζήτημα της έλλειψης εργατικού δυναμικού με αυτή την έκθεση. Ε, ενώ ταυτόχρονα όμως υπάρχει και τεράστια τεράστιε ικανότητε επαγγελματικέ οι οποίε δεν αξιοποιούνται γιατί υπάρχει και υψηλή ανεργία. Από τη μία λοιπόν πλευρά έχουμε έλλειψη εργατικού δυναμικού και ταυτόχρονα έχουμε και υψηλά ποσοστά ανεργία, ειδικότερα ανεργία των νέων, κυρίω στι νότιε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μετά έχουμε και ε, πολλές ε, περιπτώσεις ε, σύνταξη συνταξιοδότηση που αποτελεί και αυτό ένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε προσπάθειες έτσι ώστε να ενισχύσουμε, να διευκολύνουμε, να ενοποιήσουμε τους κανόνες σε ό,τι αφορά την κινητικότητα των εργαζόμενων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δεύτερο ζήτημα που θέλω να ε, υπογραμμίσουμε είναι ότι υπάρχει με ένα σημαντικό αριθμό ανθρώπων οι οποίοι ήδη διαμένουν νόμιμα εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οποίοι έχουν επαγγελματικέ δεξιότητε, ε, οι οποίε ωστόσο δεν αξιοποιούνται σε ε, μεγάλο βαθμό και δεν αξιοποιούνται αποτελεσματικά. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι αναμένουν να λάβουν, για παράδειγμα, άσυλο, άλλοι οι οποίοι αναμένουν την ε, επανένωσή του ε, με μέλη τη οικογένεια του και βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι εκείνοι, πήκο των χωρών, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά νομίμω εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωσης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τι επαγγελματικέ του δεξιότητε, να εργάζονται και με αυτόν τον τρόπο να μην επιβαρύνουν και τα ε, συστήματα κοινωνικής ασφάλειας, είτε αυτά είναι εθνικά είτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιθέτω, με αυτόν τον τρόπο δηλαδή εργαζόμενοι μπορούν να συμβάλλουν σε αυτά τα συστήματα κοινωνική ασφάλιση. Αυτά είναι λοιπόν τα δύο κυριότερα ζητήματα πάνω στα οποία θα κινηθούν οι δικέ μου τροπολογίε και αναμένω τι συζητήσει που θα ακολουθήσουν μέσα Στι στι μέρε μέρε με την εισηγήτρια. Ευχαριστώ για μία ακόμα φορά την κυρία Αραφάλης και την εισηγήτρια και ευχαριστώ και εσά, πρόεδρε. Ε, ε, η κυρία Ντούρα Φεράντη. Η κυρία Ντούρα Φεράντη τώρα για το S&D. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω ισπανικά. Ω εκπρόσωπη των σοσιαλιστών θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι σημαντικό να προχωρήσουμε σε ένα ευρωπαϊκό κοινό πλαίσιο που θα εγγυάται την προστασία και την ένταξη στην αγορά εργασία των μεταναστών που προέρχονται από τρίτε χώρε εφόσον ετούνται άσυλο ή είναι ε, πρόσφυγες ή ε, χαίρουν διεθνούς προστασίας ε, και αυτή είναι η προσέγγισή μας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά κενά, υπάρχουν πολλά εμπόδια στην πολιτική μετανάστευση και υπάρχει έλλειψη συντονισμού μεταξύ αυτών και άλλων πολιτικών κοινωνικών που σχετίζονται με την απασχόληση, δημόσιες πολιτικές που σχετίζονται με την απασχόληση, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην κατάρτιση, στην εκπαίδευση. Εδώ συνδέεται με την έλλειψη εφαρμογής των ε, διεθνών κανόνων διεθνούς δικαίου, ε, ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. χρειαζόμαστε εγγύ, κανόνες που θα εγγυώνται την, τα ίσα δικαιώματα στην αγορά Υπάρχουν οδηγίες βέβαια όπως αυτή της Blue Card, αλλά δεν εφαρμόζεται ορθώς. Θα πρέπει να τις ξαναδούμε αυτές τις οδηγίες και βεβαίως θα χρειαζόμαστε και νέα μέτρα όπως ένα νέο πλαίσιο αναγνώρισης των δεξιοτήτων που θα εγγυάται την ένταξη όλων των μεταναστών ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, ανεξάρτητα από την πορεία τους. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδέχεται τις καταχρήσεις στον εργασιακό τομέα στο έδαφος της. Και το COVID ε, ήρθε να αναδείξει μια σειρά από τέτοιου είδου καταστάσει με περιοχικού εργαζόμενου που εργάζονται παράνομα σε πολλά κράτη-μέλη τη Ένωση. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ανεχόμαστε αυτέ τι πρακτικέ. 10% του ενεργού πληθυσμού μα αποτελείται από αυτού του ανθρώπου. Η καταπολέμηση των διακρίσεων και του κατακαιρματισμού τη αγορά εργασία πρέπει να είναι προτεραιότητα για μια αγορά ενιαία που να εντάσσει. Υπάρχει μια ευκαιρία εδώ και για την κοινωνία μα αλλά και για την αγορά εργασίας και είναι κάτι που θα ενισχύσει την οικονομία στο σύνολό τη. Το να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση των υπηκών τρίτων χωρών στην αγορά εργασία μα είναι εξίσου σημαντικό όσο και για τους συμπολίτε μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό από πλευρά οικονομικής, από πλευρά δημοκρατικής και από πλευρά κοινωνική δικαιοσύνη. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Φεράντιθ και τώρα για την ομάδα Renew Κυρία Φάιλα, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Κυρία Ραφάιλα. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα εδώ, με πολλά ωφέλη για τους Ευρωπαίους, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τους Ευρωπαίους πολίτες. Και υπάρχουν βεβαίως και, υπάρχει η ηθική πλευρά. Η μετανάστευση έχει συχνά μια αρνητική χρειά, όμως οι δυνατότητες που δημιουργεί αυτή η μετανάστευση ε, δεν τονίζονται αρκετά. Η έκθεση αυτή αναφέρει ότι οι δημογραφικές αλλαγές ε, σημαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση εργαζομένων σε διάφορους τομείς της περίθαλψης, ε, της φροντίδας των, των, των ηλικιωμένων. Πρέπει η, αγορά και η ζήτηση σε ό,τι αφορά τις δεξιότητες να αντιστοιχίσουν και σε αυτό βοηθάει η μετανάστευση. Στο μέλλον θα, έρθουν πιο, θα δουλεύουν πιο πολλοί άνθρωποι μέσω της κινητικότητας ε, θα ανοίξουν και άλλο τα σύνορα και θα πάνε αλλού αυτοί οι άνθρωποι ε, και εμείς πρέπει να είμαστε να τα προλάβουμε όλα αυτά πρέπει να μπορούμε να προσελκύουμε εργαζόμενους με υψηλές δεξιότητες στην αγορά εργασίας της Ένωσης πρέπει να μπορούμε να εξασφαλίσουμε όταν προσελκύουμε τους ανθρώπους αυτούς τους νόμιμους μετανάστες θα πρέπει το σύστημά μας, η αγορά μας, η αγορά εργασίας μας να τους προστατεύει και να προστατεύει τα δικαιώματά τους και να αποφεύγουμε την εκμετάλλευση. Επίσης πρέπει να έχουμε μια ανοιχτή στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αποδοχή της νόμιμης μετανάστευσης ανθρώπων από διαφορετικά πλαίσια, από διαφορετικές ε, κουλτούρες. Ε, χρειαζόμαστε ε, προστασία των εργαζομένων που έχουν εργαστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να συμμετέχουν ισοτήμως, να προστατεύονται τα δικαιώματά τους. Ανυπομονώ βεβαίως να ακούσω τι συνεισφορές και το λοιπόν για το θέμα αυτό και να συνεισφέρω και εγώ. Ελπίζω και το μήνυμά μου προ τον εισηγητή είναι, είναι ότι η έκθεση αυτή θα είναι συμπεριληπτική. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή τύχη. Ευχαριστώ για την ID, κυρία Ωραίο, δύο λεπτά γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μα. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ραφάλσκα για αυτή την εξαιρετική έκθεση εδώ, γιατί νομίζω μας ε, ε, μας καταδεικνύει ότι ε, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ε, την δημογραφική αλλαγή χρειαζόμαστε μετανάστευση, αλλά μετανάστευση με συγκεκριμένους όρους. Αυτό είναι το σημαντικό. Αλλά πραγματικά οι συνθήκες οι οποίες θέτουμε, οι όροι που θέτουμε είναι λανθασμένοι. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι για παράδειγμα θέλουν να μεταναστεύσουν από τη Νέα Ζηλανδία, από την Αυστραλία, ακόμα και, η ε, Αυστρία για παράδειγμα είναι χώρε πολύ πιο ελκυστικέ από ότι εμεί, για παράδειγμα. Ε, κάποτε ένας ε, καγκελάριο μας πριν από 20 χρόνια, ο κύριος ε, Σιρόντερ, προσπάθησε να κινήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα ακριβώ μετανάστευση για συγκεκριμένου ανθρώπου, αλλά δεν τα κατάφερε να έχει μεγάλο αποτέλεσμα. Ε, και το Μεξικό ξεκίνησε μια αντίστοιχη πρωτοβουλία πιο πρόσφατα, αλλά κανένας τελικά δεν ανταποκρίθηκε σε αυτή την πρόσκληση. Ε, αυτό σημαίνει τι, ότι συνήθω οι άνθρωποι οι οποίοι προσέχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά κανόνα ευτοχοί και δεν έχουν τι απαραίτητε επαγγελματικέ δεξιότητε. Και επίση άλλο πρόβλημα είναι ότι έχουμε διαρροή εγκεφάλων. Δηλαδή υπάρχουν ε, ε, πολλοί δικοί μα άνθρωποι οι οποίοι εγκαταλείπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, επιστήμονε για παράδειγμα, ιατροί, πολιτικοί μηχανικοί, οι οποίοι παίρνουν και μεταναστεύουν στην Αυστραλία, οπουδήποτε αλλού, στον Καναδά, ακριβώ γιατί λαμβάνουν και ψηλότερε αμοιβέ. Άρα λοιπόν έχουμε ανθρώπου με υψηλέ επαγγελματικέ δεξιότητε που μα ε, ε, ε, εγκαταλείπουν και πολλού ανθρώπου οι οποίοι έχουν πολύ χαμηλέ δεξιότητε και προσέρχονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οποίοι δεν θα συμβάλλουν τελικά στην ευημερία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε μετανάστευση με ε, συγκεκριμένε συνθήκε, με συγκεκριμένου όρου. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε προγράμματα τα οποία θα μα καταστήσουν πιο ελκυστικού προκειμένου να προσελκύσουμε ακριβώ του κατάλληλου ανθρώπου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, λέει πρόεδρος. Τώρα η κυρία Ντεσούτερ από του πράσινου. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ε, λαμβάνω εδώ το λόγο μου του συναδέλφου Μουνιέρ Σατούρη που δεν έχει δυνατότητα να παρευρεθεί σήμερα εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν την κυρία Ραφάρισκα για ε, ε, το σχέδιο αυτό γνωμοδότηση και θα ήθελα να αναφέρω ότι η οικονομική μετανάστευση δεν αποτελεί πρόβλημα. Αντιθέτω, η εμπορία ανθρώπων είναι ε, θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε εδώ σε δυνατότητες για τους ανθρώπους οι οποίοι ε, τους μετανάστες μας ε, για να έχουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε τη δυνατότητα να μπορούν να ε, παραμένουν ε, για μεγαλύτερο διάστημα ανάλογα με την ε, συνθήκη εργασία που έχουν έτσι ώστε να προστατεύονται με τον κατάλληλο τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί λοιπόν να δώσει και μια βοήθεια εδώ παρέχοντα περισσότερε πληροφορίε για αυτού του εργαζόμενου μετανάστε και προκειμένου να μην υπάρχουν περιπτώσει εκμετάλλευση. Θα πρέπει να είναι δυνατό για όλου του μετανάστε ασχέτω ασχέτους της κατάστασή του σε ό,τι αφορά την παραμονή να έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να μπορούν να βρουν την κατάλληλη θέση εργασία και τι καλύτερε συνθήκε εργασία για εκείνου με βάση το δικό του ε, προφίλ. Η, ανθρωπιστική, η αναπτυξιακή μάλλον ε, βοήθεια θα πρέπει να είναι γενναιόδορη έτσι ώστε να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τα χάσματα ανάμεσα στο βορρά και στο νότο. Και επίση ο συνάδελφο Μονέα είπε ότι είναι σημαντικό να υπάρξουν αυτές, αυτά τα μέτρα έτσι, προκειμένου να έχουμε για παράδειγμα τι θεωρήσει, τα βίζε δηλαδή δηλαδή σε ό,τι αφορά εκείνου που αναζητούν εργασία, να έχουμε προγράμματα κινητικότητα νέων και ό,τι καθεξήν. Ε, καθεξής. Επίσης είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν ε, τα δικαιώματα των εποχιακών εργαζόμενων, ειδικότερα την, την, την πρόσβασή τους σε ε, ε, δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης, ε, δικαιώματα σε ό,τι αφορά την κατοικία ε, και ούτω καθεξής. Ε, συνάδελφος θα αποστείλει τις ε, δικές μας τροπολογίες και τα σχόλιά μας και αναμένουμε την περαιτέρω ενδιαφέρουσα συνεργασία που θα έχουμε. Ευχαριστώ και τώρα για την ΚΟΕ και ο εισηγητής ο κύριος Αρβανίτης έχει το λόγο. Παρακαλώ έχετε το λόγο. Πολύ. Ε, στο συγγνώμη που δεν είμαι κοντά σας για λόγους υγείας, αλλά την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε μαζί. Θα ήθελα να πω ότι επί τη αρχή συμφωνώ με τι ειδήσει των εκπροσώπων των Σοσιαλιστών και των Πρασίνων και θα επισημάνω μόνο δύο-τρία πράγματα και θα θέσω μια πρόταση. Είναι αναντήρητη πραγματικότητα, έτσι κι αλλιώ, πω η Ευρώπη σήμερα έχει την ανάγκη τη μετανάστευση λόγω του δημογραφικού, όπω είπαν πολλοί συνάδελφοι, αλλά και άλλων παραγόντων. Παρά στην Ευρώπη καταφεύγουν οι πίκοοι τρίτων χωρών, στην πλειοψηφία του προερχόμενοι από πολιτικά ασταθή περιβάλλοντα, ασταθή πολιτικά χώρε. Θέλω να πω ακόμα ότι ε, η ίδια συνθήκη τη Λισαβόνα προσφέρει τι νομικέ και τι θεσμικέ προποθέσει για τη μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μετανάστευση έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη τη Ευρώπη τι τελευταίε δεκαετίε. Πάνω σε αυτή την παραδοχή και αναγνώριση είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί ένα πλαίσιο για τη μετανάστευση, την νόμιμη, όχι μόνο για λόγου εργασία, οικογενειακή επανένωση σπουδών, έρευνα και γενικότερα κατάρτιση. Πάγια θέση τη αριστερά, τη ομάδα μου δηλαδή, είναι η δημιουργία ανοιχτών δρόμων υπό υποποθέσει νόμιμη μετανάστευση, με πρώτη προτεραιότητα την προστασία του αγαθού τη ανθρώπινη ζωή και παράλληλα την αποτελεσματική καταπολέμηση των διακινητών ανθρωπίνων ψυχών. Διεκδικούμε ω ομάδα πολιτική διεθνή προστασία και κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για το άσυλο, παραδοχή του αντίκτυπου τη μετανάστευση και τη κινητικότητας της ανάπτυξη. Ο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών και προέρχομαι από χώρα μεταναστών, από την Ελλάδα, συνιστά οριζόντιο θέμα στην προσέγγιση μα στο ζήτημα και δεν πρέπει ο σεβασμό αυτό να περιορίζεται στου κανόνε εισόδου και παραμονή στη χώρα υποδοχή για εργασία, αλλά και να επεκτείνεται και να καλύπτει τη συνολική ένταξη των ανθρώπων αυτών, καθώ δυστυχώ το προφίλ του μετανάστευση ακολουθεί να αποτελεί πηγή διακρίσεων στους όρους εργασίας. Πήραμε μια πρόταση. Για τους παραπάνω λόγους θα προτείνω με τροπολογία την αναθεώρηση οδηγίας για την μια κάρτα, καθώς επίσης και την υλοποίηση της πρόθεσης της Επιτροπής για την δημιουργία ανεξάρτητης αρχής για την επιθεώρηση εργασίας. Σας ευχαριστώ πολύ από την Αθήνα. Yes, thank you very much. And the last one on the list who has to take the floor would be Mr. Kosha. Mr. Kosha, we are running out of, out of time. You only have one minute. Κύριε Κώσα, έχετε μόλις ένα λεπτό για να παρέμβεστε κι εσείς. Η κυρία Κώσα, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δίνετε, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή μας, διότι το κείμενο είναι εξαιρετικά ισορροπημένο. Ε, άκουσα τους συναδέλφους και ε, βλέπω ότι έχουμε αποκλίνουσες απόψεις. Ε, βλέπουμε διαφορετικά τα ίδια θέματα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία σημεία όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να πάρει θέση. Βλέπω ότι πολλοί αναφέρονται στην αγορά εργασίας και στις ελλείψεις εκεί ως ε, μια δικαιολογία για την παράνομη μετανάστευση, λένε. Δεν μιλάμε για παράνομη μετανάστευση εμείς, μιλάμε για νόμιμη μετανάστευση. Και αυτό θέλω να το τονίσω. Επίσης, ε, πρέπει να έχουμε μια επιτυχή οικογενειακή πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μπορεί να είναι μια απάντηση στα δημογραφικά προβλήματα. Πρέπει να ενισχύσουμε την υποστήριξη των οικογενειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, νομίζω ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε την αγορά εργασία. Η ενιαία αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προστατευτεί. Να προστατεύσουμε την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Διότι παίρνονται κάποια μέτρα προστατευτισμού από διάφορα κράτη-μέλη που δημιουργούν πρόβλημα. Και δυστυχώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετείχε στην τροποποίηση κάποιων νομοθεσιών προς την αρνητική κατεύθυνση, όπως η οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων. Αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε στο μέλλον. Και τέλος, υπάρχει το θέμα της φυγής εγκεφάλων που ανέφερε ε, και ο εισηγητής. Και μια φράση ακόμα, δεν νομίζω ότι είναι σωστό μια χώρα ε, να διαθέτει οικονομικούς πόρους για την κατάρτιση, την εκπαίδευση ανθρώπων που όταν παίρνουν το πτυχίο τους, φεύγουν από τη χώρα και πάνε κάπου αλλού να εργαστούν και να πληρώνουν τους φόρους τους. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αυτό το συζήτημα στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Κώσα. Από την Κομισιόν τώρα, DG Home, η κυρία Σίλβια Γκρέκα ή ο κύριος Γκρέκα. Θέλετε να προσθέσετε κάτι σε αυτή τη συζήτηση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρακαλώ. Είναι εδώ ο κύριος Γκρέκο. Είναι συνδεδεμένος. Ναι. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή και τα αξιότιμα μέλη. Συγγνώμη κύριε Γκρέκο, σας ε, ακούμε αλλά δεν σας βλέπουμε και δεν μπορεί να υπάρξει διερμηνία αν δεν σας βλέπουμε. Ναι, συγγνώμη. Δεν ξέρω πώς να ενεργοποιήσω την κάμερα. Εξακολουθούμε να μπορούμε να σας δούμε. Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά, διότι δεν έχουμε και χρόνο αυτή τη στιγμή. Στο αριστερό μέρος της οθόνης, κύριε Γκρέκο, νομίζω μπορείτε να συνδέσετε την κάμερα. Μπορείτε να πατήσετε ένα κουμπί που υπάρχει εκεί. Ναι, συγγνώμη, από ό,τι φαίνεται δεν λειτουργεί. Θα πρέπει να προχωρήσουμε να δώσω το λόγο στην κυρία Ραφάλσκα, την εισηγήτρια, για να κλείσουμε τη συζήτηση. Κυρία Ραφάλσκα, έχετε το λόγο. Παρακαλώ, σύντομα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους ε, παρεμένους για τα σχόλια. Σίγουρα θα τα λάβω υπόψη μου στις εργασίες μου. Να αντιδράσω σε κάποια από αυτά που ακούστηκαν η κινητικότητα, παραδείγματος χάρη, των εργαζομένων. Βεβαίως, και είναι μια σημαντική πτυχή, υπάρχει το θέμα των δεξιοτήτων, Πολλοί είπαν ότι η εκπαίδευση, η αναγνώριση των δεξιοτήτων, των προσόντων είναι σημαντική. Έγινε αναφορά επίσης της καταχρήσης. Σημειώστε ότι το αντικείμενο της έκθεσης είναι η νόμιμη μετανάστευση, έτσι, και η νόμιμη εργασία. Βεβαίως το πρόβλημα αυτό υπάρχει, σίγουρα. Έγινε αναφορά στις δημογραφικές ε, αλλαγές. Βεβαίως και υπάρχει αυτό το ζήτημα, το οποίο δεν πρόκειται ε, να εξαφανιστεί αντικαθιστώντας ε, τους εργαζόμενούς μας με μετανάστες. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Έγινε αναφορά επίσης στην οικογενειακή πολιτική και στην ενίσχυση της οικογένειας γενικότερα. Και αυτό είναι ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει. Θα πρέπει να ακολουθούν οι τροπολογίες, να τις δούμε. Θα πρέπει να κάνουμε μια σύνθεση με βάση τροπολογίες. Σας ευχαριστώ όλους πάντως για τις παρεμβάσεις σας.